Ομοσπονδία Σοσιαλιστών Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου ζητήθηκε ο κύριος ε, Σαλόμα να συμπεριληφθεί στην Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων αντικαθιστώντας τον κύριο Ατόντο. Υπάρχουν σχόλια? Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν, επομένως εγκρίνεται ο διορισμός αυτός και έτσι ολοκληρώνουμε με την ώρα των ερωτήσεων. Η συνεδρίαση της Ολομέλης θα επαναληφθεί στις 9 το βράδυ.